Αναφέρομαι στην ερμηνεία του 191, του άρθρου 191, μιας και δεν υπήρξε διαφορετική άποψη για την ερμηνεία αυτή, για τη σωστή άσκηση, την ορθή άσκηση της δημοκρατίας στο κοινοβούλιο μας, θέλω να βεβαιωθώ ότι δεν θα υπάρξει αναδρομική ισχύς και αυτό δεν θα επηρεάσει τις ενισχύει εντολές και ότι ο κανόνας αυτός θα αναφέρεται και θα ισχύσει για την ανανέωση των μελλοντικών έντολων στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας.